Συμβουλίου θα υπογράψω 7 νομικές πράξεις ε, που υπόκεινται στην, έχουν εγκριθεί από την κανονική νομοθετική διαδικασία. Οι τίτλοι αυτών των νομοθετικών πράξεων θα εμφαίνονται στα πρακτικά της σημερινής μας συνεδρίασης. Και περνάμε τώρα στην ημερήσια διάταξη αυτής της Συνόδου. Για την ημερήσια διάταξη